Goedendag collega's. Het zal eh, voor sommigen onder jullie een beetje verbazingwekkend zijn dat jullie mij... Eh, Καλησπέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Φαντάζομαι εκπλήσεστε κάποιοι βλέποντα εμένα να προεδρεύω. Κυρία Γκρέσλε, δεν μπορεί να είναι όμω μαζί μα απόψε. Και πριν τι 4 δεν θα είναι εδώ και κανεί αντιπρόεδρο. Μέχρι τότε θα προεσδρεύσω εγώ. Και γιατί είμαι και ο πρεσβύτερος, τέλο πάντων είμαι αυτός που βρίσκομαι εδώ από το 1999, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Δεν είμαι ο πρεσβύτερος σε ηλικία τουλάχιστον, πάλι καλά, αλλά σε αρχαιότητα, εδώ. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν σχόλια. Εγκρίνεται η μερσιά διάταξη. Στην ενημερωτική επιστολή Cont News βλέπετε το κλασικό καθεστώς. Επίσης ε, μεταδίδεται συνήθως ε, στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις και στο σημείο 3 πρακτικά των συνεδριάσεων τη 11η και τη 18η Ιανουαρίου. Αν δεν έχετε μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση σχόλια για τα πρακτικά αυτά, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Περνάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο σημείο τη μέσια διάταξη, ε, ουσιαστικό σημείο της διάταξης, όπου θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Βουλγαρική Προεδρία. Να καλωσορίσω την Μαρινέλα Πέτροβα. Αναπληρώτερο Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας. Ε, θα συζητήσουμε για τις συστάσεις του Συμβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή του 2016. Σας καλωσορίζω κυρία Πέτρο ε, και προτείνω να έχετε καταρχάς ε, κάποιο χρόνο για να μας παρουσιάσετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και έπειτα θα ακολουθήσει συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, συγγνώμη για τη φρικτή φωνή μου. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να μπορώ να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα για να σας παρουσιάσω τις συστάσεις του Συμβουλίου για την απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση, την εκτέλεση μάλλον του προπολογισμού για το 2016 όπως προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης. Το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην ε, διαδικασία τη απελλαγή. Είναι σημαντικό τα κονδύλια να έχουν εκτελεστεί βάσει των κανόνων και οι δαπάνε να έχουν ε, ακολουθήσει τι αρχέ τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ υιοθέτησε σύσταση να δώσει την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προπολογισμού 2016 στις 20 Φεβρουαρίου. Επίσης, ενέκρινε συστάσεις για την απαλλαγή για, τις αποκεντρωμένους, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις ε, κοινοπραξίες τις κοινέ επιχειρήσεις. Σε αυτή τη σύσταση το Συμβούλιο τονίζει μια σειρά από στοιχεία που κατά την άποψή του θα πρέπει να παρακολουθηθούν και να ακολουθηθούν από όλους τους ε, φορείς αμελητή. Από την άλλη, το Συμβούλιο καλωσορίζει το γεγονό ότι για πρώτη φορά από τότε που το δικαστήριο άρχισε να δίδει τη δίδυγλωση ασφαλείας το 1994, είναι θέμα ε, της νομιμότητας και της ε, ε, σωστής εκτέλεσης των κονδυλίων και όχι το αντίστροφο. Επιπροσθέτω, το Συμβούλιο καλωσορίζει την σταδιακή μείωση του συνολικού επίπεδου σφάλματο όπω έχει υπολογιστεί από το δικαστήριο τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, το υπολογιζόμενο επίπεδο σφάλματο ε, υπολογίζεται για τι πληρωμέ σε 3,1% και είναι πάνω από τον δείκτη αξιολόγηση του 2%. Το Συμβούλιο, λοιπόν, επαναλαμβάνει την επιθυμία του να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσει στη συστήματα οικονομική διαχείριση και στο υπολογιζόμενο επίπεδο σφάλματο σε διάφορου πολιτικού τομεί πολιτική. Πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι αυτά που επιτεύχθησαν ως τώρα και σε αυτό το πλαίσιο οδηγούν το Συμβούλιο να εκφράσει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Είναι θετικό ότι η αγορά και οι άμεσες ε, δαπάνες στήριξη στο κεφάλαιο 2 δεν επηρεάστηκαν από τα ασφάλματα υλοποίησης το 2016. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η αγορά και η άμεση στήριξη είναι τα 3 τέταρτα των δαπανών ε, υπό αυτό το κεφάλαιο, ωστόσο, υπό αυτό τον τίτλο. Ωστόσο υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει. Το Συμβούλιο καλεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις συστάσεις του δικαστηρίου. Επίσης καλεί τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσουν ε, έμφαση στην αύξηση της ποιότητας, περισσότερο από ό,τι στην ποσότητα, στα πρώτα επίπεδα ελέγχου και προκειμένου να μπορούν να ανοιχνεύσουν ε, και να διορθώσουν σφάλματα και κυρίως να τα προλάβουν. Το Συμβούλιο κυρίως τονίζει ότι οι έλεγχοι δεν είναι ανευκόστους, λαμβάνοντας υπόψη το περίπλοκο των πολιτικών και των προγραμμάτων. Ε, Κατά συνέπεια, πρέπει να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ του κινδύνου σφάλματο και του κόστου ελέγχου και ορκωτών ελέγχων, επικεντρωνόμενοι σε καλύτερου ελέγχου περισσότερο σε ποσότητα, σε αριθμό, μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων. Η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη διόρθωση. Η Επιτροπή ε, τονίζει ότι χρειάζονται μέτρα πρόληψη, όπω η διακοπή και η αναστολή πληρωμών, βάσει των ισχυρών κανόνων. Το Συμβούλιο επίση τονίζει την ανάγκη να συνεχίσουν να γίνονται οικονομικέ διορθώσει και ανακτήσει με αυστηρότητα βάσει των ε, ισχυών των κανόνων, προκειμένου να προστατευτεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Υπό αυτήν την έννοια πρέπει να πούμε επίση ότι το Συμβούλιο εκφράζει την δυσαρέσκειά του που δεν χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί τι διαθέσιμε πληροφορίε για να προλάβουν, να ανοιχνεύσουν και να διορθώσουν ένα μεγάλο αριθμό σφαλμάτων. Αυτό θα είχε μειώσει σημαντικά το υπολογιζόμενο επίπεδο σφάλματο, ώστε να φτάσουμε κοντά στο πραγματικό ε, όριο σε όλα τα κεφάλαια δαπανών. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ιδιότητα του πολίτη, την ε, υπηκότητα, για πρώτη φορά το Συμβούλιο καλωσορίζει το γεγονός ότι το δικαστήριο αφιέρωσε στην έκθεσή του ένα ειδικό κεφάλαιο στο θέμα αυτό. Ενθαρρύνει το δικαστήριο να συνεχίσει αυτό τον έλεγχο παρακολουθώντα όλο αυτό το πεδίο και κοιτάζοντα το επίπεδο σφάλματο, τι συστάσει και τι πληροφορίε για τι επιδόσει. Επιπλέον, το Συμβούλιο τονίζει ότι οι δαπάνε στον τομέα αυτό έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίω λόγω των πολιτικών μετανάστευση. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να αυξηθεί η ένταση των ελέγχων. Θα ήθελα να προτείνω στους ευρωβουλευτές ε, η ε, Επιτροπή σας να ενθαρρύνει επίσης το δικαστήριο να συνεχίσει τους ε, ελέγχους για αυτόν τον τίτλο. Τέλο, το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τι αδυναμίες που έχει βρει και το δικαστήριο, εφαρμόζοντα τα συστήματα ελέγχου που ισχύουν στου τομεί τη μετανάστευση και τη ασφάλεια. Και τώρα να στραφώ στην ε, δημοσιονομική και την οικονομική διαχείριση και την προβλεψιμότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Το χάσμα μεταξύ των εγκεκριμένων και των ε, ε, πληρωμών που χρησιμοποιήθηκαν, των δεσμεύσεων πληρωμών που χρησιμοποιήθηκαν, αυξήθηκε το 2016 και το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του γεγονότος. Αναγνωρίζεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη πίεση τα επόμενα χρόνια στις πληρωμές. Ε, για αυτό το λόγο το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προλάβει αυτή την εξέλιξη με μια τακτική ε, εκταμείευση πληρωμών προκειμένου να μην υπάρξουν ελλείψεις και κενά. Το Συμβούλιο παρατηρεί ότι τα ΡΑΛ είναι σε αύξησης και εκφράζει την ανάγκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό και να ελέγχει την διαφορά μεταξύ δεσμεύσεων και ε, των ε, πληρωμών που έχουν αναλυθεί. Ε, μια άλλη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη δυσονομική έκθεση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, με τις μακροπρόθεσμες, ε, με, τις μακρο, με τα μακροπρόθεσμα στοιχεία παθητικού, τις εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις. Υπ' αυτήν την έννοια το Συμβούλιο ε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις και το σχετικό οικονομικό κίνδυνο. Τέλος, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εντείνει την διαφάνεια, απλότητα και λογοδοσία των εργαλείων Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Και ένα τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι οι επιδόσεις. Το να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα και να επικεντρωθούμε στις επιδόσεις είναι ε, ύψης της σημασίας, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχία και της έλλειψης πόρων. Το Συμβούλιο εκτιμά το έργο του δικαστηρίου προκειμένου να αποτιμήσει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να κάνει μια ετήσια αξιολόγηση τη καστή οικονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε το δικαστήριο να συνεχίσει να δίνει έμφαση στις, στο σκέλος των επιδόσεων στις μελλοντικέ αιτήσεις εκθέσεις του. Το Συμβούλιο συμφωνεί με την σύσταση του δικαστηρίου να παρακολουθήσει και να ευθυγραμμίσει την υποβολή εκθέσεων για τις επιδόσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο είναι συνεκτικοί οι στόχοι και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στις δηλώσεις του προγράμματος και στις διάφορες δράσεις των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, βελτιώνει διαρκώς τη δυνατότητα υποβολής εκθέσεων στο σκέλο των επιδόσεων, με ποιότητα των πληροφοριών, αύξηση της διαφάνειας, του εύληπτου και τη φιλικότητας προ το χρήστη. Όσο πιο ισόρροπε είναι σε αυτές οι εκθέσει, τόσο καλύτερα θα γνωρίζουμε τι παρελθούσε επιδόσει. Αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με περισσότερε πληροφορίε και θετικά παραδείγματα, αλλά και με επικέντρωση στι βασικέ προκλήσει για να επιτευχθούν αποτελέσματα, να σημειωθούν τα κενά και ε, τα σημεία αποτυχία. Το Συμβούλιο τονίζει ότι η ενίσχυση του πλαισίου επιδόσεων θα πρέπει να σέβεται την ισορροπία μεταξύ κόστους και ωφελίας από την καταγραφή των πληροφοριών επίδοσης. Θα πρέπει με τους ανάλογους δείκτες να έχουμε τα σωστά δεδομένα για να αποφύγουμε το περιττό γραφειοκρατικό άχθος. Ο αριθμός των στόχων και δικτών πρέπει να εξορθολογιστεί και τελικώς να μειωθεί. Κυρίες και κύριοι, αφού τα είπα όλα αυτά, δεν μπορώ παρά να συμπεράνω ότι το επίπεδο σφάλματος που έχει υπολογίσει το ελεγκτικό συνέδριο είναι αποτέλεσμα των μέτρων ε, ε, δεν είναι αποτέλεσμα των μέτρων για την απάτη, την ε, αναποτελεσματικότητα ή την κατασπατάληση των κονδυλίων αυτή καθεαυτή. Θα πρέπει όλοι οι θεσμοί και οι εμπλεκόμενοι να χρησιμοποιούν καλύτερα τα κονδύλια με μεγαλύτερη προσοχή και να ακολουθούν τι σχετικέ απαιτήσει. Α βεβαιωθούμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, αξιοποιούνται για να επιτύχουμε αποτελέσματα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα προ του Ευρωπαίου πολίτε και φορολογουμένου ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται με τρόπο υπεύθυνο και ότι υπάρχει πλήρη λογοδοσία. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. inleiding. Ευχαριστώ πολύ, Σας κυρία ευχαριστώ. Υπουργέ. Έχω εδώ γραμμένο τον κύριο Βοητσεχόφσκι και τον κύριο Σάραβαμα. Υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Εδώ εσείς σας σημειώνω. Και παρακαλώ να εγγραφεί και το δικό μου όνομα. Ο κύριος Ζντεχόφσκι. Κανονικά βέβαια λαμβάνει το λόγο ο συντονιστής κύριε Πρόεδρε, αλλά με, για μεγάλη μου χαρά μου δώσατε εμένα πρώτο το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Στην παρέμβασή σας, κύριε Υπουργέ, είπατε θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικτών και των στόχων. Καμιά φορά όμως εμείς βρίσκουμε ότι τα προγράμματα είναι υπερβολικά πολλά και λίγα από αυτά αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Εμείς θα προτιμούσαμε λιγότερα προγράμματα τα οποία να μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα. Γι' αυτό και τοποθετηθήκαμε και με ειδική έκθεση σχετικά με το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα αυτό το greening είναι ένα ε, παράδειγμα μιας καλής πρόθεσης που ωστόσο δεν οδηγεί στα αποθούμενα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα θέλαμε πολύ το Συμβούλιο να προβληματιστεί περισσότερο για το θέμα αυτό, να ασχοληθεί περισσότερο και να υποστηρίξει περισσότερο την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι όπου κάτι δεν λειτουργεί πρέπει να το αντιμετωπίζουμε λογικά και να το τροποποιούμε, να μην το αφήνουμε απλώς να συνεχίζει να λειτουργεί. Μιλήσατε και για το ποσοστό σφάλματος και για τους δείκτες. Το ποσοστό σφάλματος, ωστόσο κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο σημαντικό. Πολλοί μιλούν για το ποσοστό σφάλματος. Αλλά τέλος πάντων τι είναι το ποσοστό σφάλματος. Το ποσοστό σφάλματος εξαρτάται από το εάν η χώρα μέλος είναι διατεθειμένη να κοινοποιήσει τα σφάλματα στις Βρυξέλλες ή όχι. Αν τώρα στη Βουλγαρία ληφθεί μια απόφαση για να, δείξει, για να δείξει ας πούμε η χώρα αυτή ότι τα πάει μια χαρά, δεν ε, κοινοποιεί τα, ε, τον αριθμό των σφαλμάτων και άρα θεωρούν οι Βρυξέλλες ότι ε, το ποσοστό σφάλματος στη Βουλγαρία είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ε, εννοώ δηλαδή ότι εξαρτάται από την προσέγγιση της κάθε χώρας μέλους. Υπάρχουν, προβλήματα, τα, ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα παρόλο που στα χαρτιά έχουν χαμηλότερο ποσοστό σφάλμα από την Τσεχία τη Βουλγαρία ή και τη Ρουμανία. Γι' αυτό νομίζω χρειάζεται να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση για το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό και η Βουλγαρία να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή, άλλωστε το υποσχέθηκε η ίδια υπουργό. Και να εξορθολογήσουμε και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την εργασία μας. Αυτό θα αποδώσει πραγματικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές χώρες ακόμα και ισχυρές λεγόμενες χώρες μέλη, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να ασχοληθούν με τις ε, περιπτώσεις απατών. Υπάρχουν εκθέσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απατών, της Όλαφ. Στην Τσεχία είχαμε μια σχετική υπόθεση όπου τέθηκε το ερώτημα αν πρέπει να δημοσιευτεί η σχετική έκθεση, όχι και μάλιστα πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές και ούτω καθεξής. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη προσέγγιση. Δεν πρέπει να εξετάσουμε ανά πάσα περίπτωση αν πρόκειται να γίνουν εκλογές σε μια συγκεκριμένη χώρα. Να επιλέξουμε, να υιοθετήσουμε μια ενιαία στάση και να κοινοποιούμε το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας εδώ να δεχτείτε την κριτική μας, διότι αυτή είναι η δουλειά μας εν τέλει. Αλλά πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας. Ο κύριος Σάρβαμα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ. Ε, σημαίνει πολλά για μας. Και από την άλλη μεριά βέβαια δεν θα πρέπει κάτι τέτοιο να είναι και τόσο σπάνιο, εξαιρετικό φαινόμενο. Ωστόσο, συγχαίρω την Βουλγαρική Προεδρία για την ενεργό συμμετοχή της εργασία μας. Σημαντικό λοιπόν και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είμαστε υπέρ της προσέγγισης της βασισμένης ε, στην αξιολόγηση κινδύνου, risk-based, ζητούμε καλύτερη απόδοση, αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού, ε, δημοσιονομικές διορθώσεις, περισσότερη διαφάνεια, απλούστευση Τώρα ίσως ας πούμε σε μια πανεπιστημιακού χαρακτήρα συζήτηση θα λέγαμε ότι είναι απολύτω κατάλληλη χρονική στιγμή για να εφαρμοστούν ορισμένα από αυτά, αλλά έχουμε μπροστά μας το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα το ΠΔΠ μετά Πού τοποθετείτε το Συμβούλιο. Δεν αναμένω να μας πείτε την πραγματική αλήθεια, αλλά ας το πω διαφορετικά. αν δεν υπάρχει πραγματικά γνήσιο ανοιχτό πνεύμα σχετικά, βρισκόμαστε σε μεγάλη δυσκολία. Όλοι, οι οι πόροι, έχουμε ανοιχτό πνεύμα απέναντι στους ίδιους πόρους. Και αν όχι, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις το Κοινοβούλιο λαμβάνει μια σκληρή, ξεκάθαρη θέση για την περίοδο μετά τη Βρετανική αποχώρηση, το Brexit. Τα είπαμε αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα πούμε και στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ακούσαμε διευθυντήριες γραμμέ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο αυτό μας ε, ενδιαφέρει όλους. Ευχαριστώ ε, η κυρία Κάπελ, ευχαριστώ. Είμαι η συγγήτρια για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως για το 2016. Ποσοστό φάρματο της τάξης του 1,7% το οποίο είναι ικανοποιητικό διότι είναι κάτω από το κατόφλιο του 2% που είναι το κατόφλιο στόχος. Η δε δήλωση αξιοπιστίας του ελεγκτικού συνεδρίου δόθηκε και σε ό,τι αφορά την νομιμότητα των διαδικασιών διαπιστώσαμε μάλιστα μείωση κατά 3,3% των δαπανών το 2016. Συμφωνώ με τα όσα δηλώσατε, ιδίω σε ό,τι αφορά τα διάφορα σχέδια, project και τη χρηματοδότησή τους, ότι πρέπει δηλαδή να διασφαλίζεται προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με βεβαίω ε, βασική αρχή την βελτιωμένη νομοθεσία και στα project αλλά και για το έργο των οργανισμών και των ταμείων για να αντιμετωπίζονται ορθά οι δεδομένες ανάγκες. Ευχαρίστως, μαζί με τους άλλους συνεισηγητές, θα λάβω υπόψη τις συστάσεις σας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως. Για τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε έχουμε προθεσμία μέχρι τις 11 Τρίτου. Αντελήφθην ότι δηλώσατε ικανοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής. Και όπως είπα, τις προτάσεις σας θα τις λάβουμε υπόψη, σας, υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νοβακόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τη απευθύνω συγχαρητήρια για την εργασία της. Θα συμφωνήσω με τον παρακαθήμενο Σάρβαμα ότι όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες κάθεται ένας ελέφαντας μέσα στην αίθουσα και αυτό θα είναι η επόμενη πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ θα πω και κάτι ακόμη. Λίγες ημέρες μετά από για την ε, απαλλαγή και τα διδάγματα που θα συναγάγουμε από αυτό θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατό, στον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο θα... Τι νομίζετε για τις ε, simplified cost options ώστε για να μειωθεί ε, το ε, ποσοστό σφάλματος και ιδίως ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ και εσάς βεβαίως κυρία Υπουργέ, κύριο Σέλερ, για την συζήτηση για την απαλλαγή 2016. Είμαι εισηγητής για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm. Η θετική σας εκτίμηση, την οποία μας εξηγήσατε μας βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνους. Όμως, πώς η συζήτηση στο Συμβούλιο, διότι λάβαμε προ λίγων ημερών επιστολή από δύο υπουργούς οικονομικών, Σουηδίας, Ολλανδίας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν διαφορετικά στην ψηφοφορία και παραπονούνται ότι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από δεκαετιών εξακολουθούν να μην γίνονται σεβαστοί. Ότι τα ποσοστά σφάλματος είναι ιδιαίτερως υψηλά. Ενώ εμείς είδαμε να μειώνονται τα τελευταία χρόνια και να ελαχιστοποιούνται. Και οι οποίοι οι υπουργοί ζητούν απαλλαγή για τον προϋπολογισμό πιο, ε, με μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται να επιτυγχάνουν το σκοπό τους. Τι άποψη έχετε για τις μομφές αυτές που προβάλλονται, όπως είπα, από δύο χώρες μέλη. Και ίσως να μην το λένε τόσο ρητά, αλλά πάντως στρέφονται κατά των διαφθορτικών ταμείων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Διότι μιλούν για νούμερα τα οποία συνδέονται ακριβώς με τα διαφθορτικά ταμεία. Δεν μιλούν καθόλου, για παράδειγμα, για τη γεωργία. ενώ εγώ νομίζω ότι χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση στις πληρωμές εκεί. Δυστυχώς, κατά την απορρόφηση των διαφθορτικών ταμείων σε πολλές χώρες, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τις περιόδους χρηματοδότησης. Άρα θα χρειαστούν κάποιες έξτρα προσπάθειες από κάποιες χώρες μέλη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που βάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Όπως είπαν άλλοι συναδελφοί μου πριν, θα πρέπει και μετά το 2060 να μιλήσουμε και για το μετά. Για αυτό, από την περίοδο αυτή. μάλλον εννοεί το 2016. Πώς θα διαμορφωθεί δηλαδή στο μέλλον ο προπολογισμό. Εκφράζουν πολύ τον φόβο ότι η πολιτική της συνοχής και τα διαφορετικά ταμεία κάπου θα χαθούν, δηλαδή θα λαιλατηθούν. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον μας, διότι η πολιτική της συνοχής είναι από τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν πολλά επίπεδα της ευρωπαϊκής πολιτικής ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι και το περιφερειακό. Και ακόμα και αν δεν φτάνουμε στο ποσοστό του 2% χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις. Και οι αποδόσεις που έχουν επιτευχθεί από τα διορθωτικά ταμεία ως μέσο επενδύσεων σε χώρες μέλη στην απασχόληση χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και για απασχόληση και για ανάπτυξη για να ξεπεραστεί ό,τι έχει μείνει από την... Ευχαριστώ πολύ. Eh, Σα ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω. Έχω εγγραφεί στον κατάλογο των μιλητών. Κυρία Πέτροβα, έχω και εγώ κάποια ερωτήματα. Τα αντιμετωπίζουν κάπως ε, ως ρουτίνα ε, από το Συμβούλιο όλα αυτά. Διαβάζουν τα έγγραφα για την απαλλαγή. Εμείς όταν θέλουμε να αποφανθούμε για την απαλλαγή, μιλούμε με τους ε, οργανισμούς αυτούς και με έναν από αυτούς τον νεάζω ενδεχόμενα σφάλματα σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, το Συμβούλιο τα αντιμετωπίζει όλοι και είπε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι για πολλά χρόνια αναβάλλουν και τότε είχαμε καταθέσει έναν επίσημο έγγραφο, έναν non-paper, για να δούμε τις διάφορες σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών και πώς θα έπρεπε να γίνεται αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών. Ένα έγγραφο το οποίο, μεταξύ των διαθεσμικών οργάνων, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δεν συνέβη όμως αυτό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν έχετε πληροφορίες και γνωρίζετε κάποιο χρονοδιάγραμμα εντό του οποίο θα μπορούσε να ενήλικοι να συμπεριφερόμαστε ένας προς ε, τον άλλο. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής, συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε ο συνάδελφος Τσέλερ. Δύο κράτη-μέλη, Ολλανδία, Σουηδία, ασκούν ε, επικρίσει, θέλουν δε μία δυσέλιδη επιστολή, δηλαδή δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένες από την περιθωριακή βελτίωση αυτή, την οριακή βελτίωση των ποσοστού σφάλματος. Αν αυτό δεν το συσχετίσουμε με το τι γίνεται με τις απαλλαγές του ελεγκτικού συνεδρίου που πολλές φορές λέει ότι τα ποσοστά σάλματος τα γνώριζαν τα κράτη-μέλη. Άρα έχουν συνυπευθυνότητα. Είναι συνυπεύθυνα μάλλον για αυτή ε, την κατάσταση. Όταν λοιπόν στο Συμβούλιο συνέρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών δεν θα πρέπει να το συζητήσουν κάποια στιγμή. Να το γνωρίζει τελευταίο ερώτημα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών χωρίς απαλλαγής Έχουμε τον ΙΣΙΝΔΙΟ, τον προϋπολισμό και το να έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών χορήγησης απαλλαγής. Έχουμε τον ΙΣΙΝΔΙΟ, τον προϋπολισμό και τον να ξεκάθαρη. Στην Επιτροπή μας το συζητήσαμε, το θέμα της διαδικασίας και με το ελεγκτικό συνέδριο. Το συζητούμε εδώ και, και ετήσια απαλλαγή θα μπορούσε να γίνει λίγο νωρίτερα και θα προσπαθήσει να καταθέσει κάποιες ε, προτάσεις αντί να πηγαίνουμε τον Νοέμβριο, Οκτώβριο, ίσως και Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να συμφωνήσετε από πλευρά Συμφουλίου για να γίνεται απαλλαγή στο έτος νησινένα. Θέλει κανείς, στρέφομαι προς αδέλφους, άρα αφού κανείς δεν θέλει το λόγο, κυρία Πέτροβα, παρακαλώ πείτε μας τις απόψεις για τις ερωτήσεις. Thank you. Uh, first, thank you for... Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον και για τα πολλά ερωτήματα που δεν είναι και τόσο εύκολα. Θα προσπαθήσω όμως να τα απαντήσω για το 2% ιδέως στην πολιτική συνοχή και στην ανάπτυξη της υπαίθρου όμως. Αν βγάλουμε τις άμεσες πληρωμές. Όμως θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι υπάρχει σταδιακή βελτίωση πρόσφατα στους τομείς πολιτικής αυτούς και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Το Συμβούλιο γνωρίζει ότι τα κράτη-μέλη και οι διχρηστικές αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στις εταιρικά της διαδικασίας, επειδή όμως είναι άκρος πολύπλοκες αυτές, είναι ότι δυσκολεύονται ιδιαιτέρως. Άρα, η απλούστευση των σχετικούς Άρα ο καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων θα μειώσει το διοικητικό άχθος, άρα και τον κίνδυνο σφάλματος και θα επιτρέψει ελέγχους Ναι, πράγματι το είπα αυτό σήμερα. Αλλά δείτε τα ποσοστά σφάλματων πολλών χωρών. Εμείς τα τελευταία τέσσερα χρόνια τουλάχιστον ε, που τα κοιτούμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ε, γελάω βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη, αλλά αναφέρουν ε, ελάχιστα σφάλματα. Και οι αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τελείως διαφορετικές σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η απόψη μου, μπορείτε να το δείτε, να το εξετάσετε. Find a solution how to do it better. Αν συμφωνήσετε, καλό θα ήταν να δείτε αν μπορεί να βρεθεί και κάποια λύση για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Κυρία Πετρόβα, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα ε, του ενωσιακού προϋπολογισμού, νομίζω μια ερώτηση που σχετίστηκε και με την ερώτηση του κ. Νοβάκοφα θα πρέπει να εστιάζουμε λίγο περισσότερο στις επιδόσεις και όχι στα σφάλματα. Όπως είπα, το Συμβούλιο χαιρετίζει το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου ε, σε ό,τι αφορά ε, την ανάλυση των επιδόσεων. Ένα στέρεο πλαίσιο επιδόσεων συνεισφέρει στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και στη σωστή αξιολόγηση της λειτουργίας των προγραμμάτων υπό το τρέχον επιδελταπή η σύσταση του Συμβουλίου ουσιαστικά παραλαμβάνει και τη σύσταση του Ελεκτικού συνεδρίου να υπάρχει εξορθολογισμό τη αναφορά των επιδόσεων. Τονίζουμε όμω εμεί ότι αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ισορροπημένο. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτιστούν δείκτε ώστε να δίδονται σημαντικά δεδομένα χωρίς όμως να αυξάνεται το διοικητικό άρθρος Θέλουμε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ της καλή απόδοσης και ενός χαμηλού ποσοστού σφάλματος. Σε ό,τι αφορά το πολιετές μουσιονικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο, όπως γνωρίζετε, εξακολουθούμε να μην έχουμε την πρόταση της Κομισιόν. Συζητήσεις γίνονται προς το παρόν και δημοσιοποιήσει την πρότασή της Κομισιόν, οπότε θα ξεκινήσουμε την ανάλυση των προτάσεων ελπίζω να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς για να διευκολύνουμε και την Αυστριακή Προεδρία που έπεται. Ορίστε. Δεν θα μας δώσετε ούτε ένα το σοδά, κάτι, μια πληροφορία. Εκτός μικροφώνου, Υπουργός. That... Όχι, ρωτούσα. Δεν θα μας δώσετε τίποτα. Ε, με τόσο δούλα πληροφορία, κάτι κύριε Πέτροβο. Να σας δώσω τη δική μας. Έχουμε όμως και τον προσανατολισμό και την καθοδήγηση που μας έδωσαν οι αρχηγοί κατοικίες. Αλλά το σημαντικό είναι πρώτα να συζητηθούν οι προτεραιότητες ε, και πώς ε, μπορούν να καλυφθούν αυτές από τον ενωσιακό προπολογισμό. Και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για τα επίπεδα πάνω. Κύριε Σάραφα, α, τώρα κατάλαβα τι έπρεπε να σας χαρωτήσει και θα το αναδιατυπώσω το ερώτημα. Πιστεύετε ως ασκούσα την Προεδρία πως θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε τις πραγματικές προτεραιότητες. Τι πρέπει να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και μόνο μετά να συζητήσουμε τα περί κόστους και μόνο μετά να δούμε προτεραιότητες. Ποια είναι τα καθήκοντα, ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι προτεραιότητες είναι σημαντικέ. Είμαστε από το Συμβούλιο όμω των Υπουργών Οικονομικών, άρα έχουμε και του δημοσιονομικού περιορισμού. Δεν μπορούμε να συστήσουμε μόνο ανοιχτά τι προτεραιότητε. Μου είπε και ο Χάνς, και αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε ε, γιατί υπάρχουν θετικέ προτεραιότητε, αλλά υπάρχουν και αρνητικέ προτεραιότητε. Σίγουρα είναι η πρώτη φάση, η γεράρχηση των προτεραιοτήτων πρέπει όμω και του δημοσιονομικού περιορισμού να του έχουμε υπόψη. Και χρονικού περιορισμού. Και διαβάζοντα τη σχετική δισιογραφία βλέπω ότι συζήτησαν περί προτεραιοτήτων και όχι, μάλλον αν εμείς μιλούμε περί προτεραιοτήτων και όχι περί χρημάτων, σε δύο χρόνια ακόμα βήμα σημειωτών θα κάνουμε. Διότι οι απόψεις διήστανται. Δηλαδή περίπου πού βρίσκονται οι δημοσιονομικές μας δυνατότητες και μετά να έλθουμε να βάλουμε προτεραιότητες. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τροφοδοτείται κυρίως από τις φορές των χωρών μελών. Θα το ξεπεράσουν είναι διατεθειμένες να τροφοδοτήσουν τον προπολογισμό με λίγο περισσότερο από αυτό. Εάν η προσπάθειά τους είναι να διατηρήσουν τις φορές των ευρωπαϊκό προπολογισμό όσο το δυνατόν χαμηλότερες, ε, αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ωστόσο, η διάσκεψη κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας δεν έδωσε πολλές ελπίδες. Και τώρα βέβαια εσείς καλείστε να σηκώσετε το βάρος αυτό και να εξηγήσετε τα σχετικά. Γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τη δική σας φωνή, αν είστε διατεθειμένοι, η Προεδρία σας δηλαδή, η οποία έχει μπροστά ακόμα μερικούς μήνες, η αιτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε υπερβαίνει η προσπάθεια αυτή το χρονικό σημείο των ευρωεκλογών και μέχρι όταν αναλάβει νέα επιτροπή και να είναι σε θέση να δράσει κτλ. θα έχουμε ακτική ανάγκη να βιαστούμε λίγο. Η Κομισιόν τουλάχιστον υπεσχέθη ότι θα καταθέσει πρόταση ήδη τον Μάιο. Αυτό βεβαίως εμπίπτει μέσα στην δική σας Προεδρία. Και θα πρέπει να υπενθυμίσετε στους ομολόγους σας ε, υπουργούς ότι είναι η σειρά τους μετά να αναλάβουν δράση και ότι χρειάζονται κάποιοι συμβιβασμοί στη βάση των διαθεσίμων και ότι στη βάση των διαθεσίμων αυτών ποντιλίων, πόρων θα πρέπει να μπουν και προτεραιότητες. Δεν είναι και πολλά. Πόσα θα δώσουμε στη γεωργία, πόσα θα δώσουμε στην πολιτική συνοχής ως διαρθρωτική πολιτική για όλες τις περιφέρειες. Θα υπάρξει ειδική γραμμή του προπολογισμού για τη μετανάστευση και τι κάνουμε με την πολιτική ανάπτυξη και πόσο θα μας κοστίσει η έρευνα. Αυτά είναι. Πέντε ερωτήματα είναι αυτά, πρέπει να απαντηθούν. Όμως δεν έχετε την πολυτέλεια του άπειρου χρόνου, διότι εξήγησα προηγουμένως και ποιες είναι οι προθεσμίες. Και νομίζω ότι η φιλοδοξία σας θα πρέπει να είναι μέχρι τον επόμενο Απρίλη, του επόμενου χρόνου, να έχετε προχωρήσει τα πράγματα αρκετά και εδώ η Προεδρία σας καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ και για αυτήν την ε, ερώτηση. Η Προεδρία μας είναι η πρώτη από το τρίο όσων θα ασχοληθούν με το πουδουπού. Εάν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για να ολοκληρώσουμε όμως τις διαπραγματεύσεις εντός της θητείας αυτή του Κοινοβουλίου πριν τι εκλογέ. Ωστόσο, η πρόταση έρχεται στο τέλο τη προεδρία μα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε, να οργανωθούμε στο επίπεδο των αρχικών δηλώσεων τι ουσιαστικέ συζητήσει και διαπραγματεύσεις θα τι ξεκινήσει η Αυστριακή Προεδρία. Και έχουμε συζητήσει εντατικά με του συναδέλφου μα από την Αυστριακή και τη Ρουμάνικη Προεδρία. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία μαζί τους και θελήσαμε να είμαστε καταρχάς ρεαλιστές, κατά πρώτον ρεαλιστές και έπειτα φιλόδοξοι. Πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας και για τις άλλες χώρες. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε στο υπόλοιπο τμήμα της Προεδρίας μας. Είναι να ενισχύσουμε δεύτερον. Τα, οι οροφές στο συνολικό ποσό του Πουδουπού και τρίτον, ε, το σωστό χρονικό σημείο, η σωστή συγκυρία. Υπήρξαν βεβαίω διαφωνίε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανεί. Στην προστασία, την ασφάλεια και τη μετανάστευση και άλλη στη συνοχή παρά τι περικοπέ. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ψηλότερα επίπεδα δαπανών. Αυτά πρέπει να συζητηθούν εν Δεν πάμε στις άλλες ερωτήσεις. κυρία Κάπελ. Α, ναι, κυρία Τσέλερ, που έλεγαν ότι καλωσορίζουν τις αντικές εξελίξεις στο ποσοστό σφάλματος, αλλά θεωρούσαν ότι αυτό δεν είναι αρκετό ακόμη για να είναι πλήρως θετική και να συμφωνήσουν με τη σύσταση. Δικαίωμά του είναι να το κάνουν. Η πλειοψηφία του, του Συμβουλίου ψηφίζει. Εξού και προκύπτουν οι συστάσεις αναρνητικά. Ναι, αλλά έγινε συζήτηση με τα υπόλοιπα κατημέλη. Διαφωνήσατε, ε, δεν συζητήθηκε καν. Ο πρέπει να αλλάξει ξεκινώντας από την ε, εθνική διάσταση ώστε το τελεκτικό συνέδριο να ξεκινήσει με την προετοιμασία, να γίνει μετά συζήτηση στο Συμβούλιο και να καταλήξουμε στη σύσταση. Γι' αυτό είναι κάπως δύσκολο να γίνει. Είπατε κάτι για ένα non-paper. Το οποίο πήγε στο Κορεπέρ. Το οποίο έδωσε εντολή διαπραγματευτική στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για να δουν ποιες είναι οι διάφορες on on on the. the How much time will that take? As soon as possible. I don't know because they are still discussing. Δεν ξέρω γιατί συζητάνε ακόμα. Δεν μπορώ να σας πω χρόνο. Όλαφ κατά εάζω. Να ξεκινήσουμε με την ε, υπόθεση ότι όλα θα Να ε, ακόμη ε, κάνει έρευνες για τον οργανισμό, για το άσυλο και αν συγκεντρωθούν, μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, θα δει το Συμβούλιο πώς θα τοποθετηθεί για τον ελόγο οργανισμό. Μπορεί να προκύψει αναθεώρηση τροποποίηση μεταρρύθμιση. για τους οργανισμούς. Το Συμβούλιο βασίζεται στους κανόνες που ισχύουν από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς που ορίζουν το πώς χειρίζονται τους λογαριασμούς στο ελεκτικό συνέδριο και όλοι οι σχετικοί φορείς. Σημειώνουμε όσα είπατε για την Όλαφ και τους άλλους οργανισμούς. Και αυτή είναι η αρχή που ακολουθεί το Συμβούλιο. Δεν μπορώ να πω να είναι επίσημη, επίσημη αυτή η διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει άλλη διαφορετική μεταχείριση για τους επιμέρους οργανισμούς. Ναι, και η κυρία Κάπελ έκανε μια ερώτηση. Και ο κύριος Νοβακόφσκι. Και ο κύριος Τσέλερ θέλει και το λόγο. Mr. Τσέλερ. Ο κύριος Τσέλερ. Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, γνωρίζω ότι δεν είστε πραγματικά η, ας πούμε, η σωστή συνομιλήτρια για να κάνω την ερώτηση αυτή. Γνωρίζω ότι είστε πολύ θετικά τοποθετημένοι απέναντι στα δικαιώματα συναπόφαση του Κοινοβουλίου και όχι μόνο προσωπικά αλλά γενικότερα. Τα καταφέρουν με αυτή τη ρύθμιση με τι προθεσμίε ώστε μέχρι το 2019, μέχρι δηλαδή τι ευρωεκλογέ, να μην καταλήξουν σε συμπέρασμα, σε κανένα αποτέλεσμα. Και να μιλήσει και αυτό θα συμβεί και με το επόμενο κοινοβούλιο. Και τα μέλη του Συμβουλίου ας έχουν υπόψη την θέληση και θα επιμείνει να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία την θέληση και θα επιμείνει να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Το σημειώνω αυτό που είπατε και θα μεταφέρω το μήνυμά σας στους συναδέλφους μου. Για το EDF είναι άντι η υπόθεση του Συμβουλίου αυτή, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτηση σας αυτή. Η τελική ερώτηση είναι του κ. Νοβακόφ, υπόδοση και για τα ποσοστά σφάλματος η απλούστευση και η αξιοπιστία της διαδικασίας πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Λόγω της θέσεως της Σουηδίας, ε, της Ολλανδίας αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου έκανα και εγώ μια ερώτηση, σημειώνει ο Μπαρτ Στάς, σχετικά με το γεγονός ότι το ECA εδώ και κάποια χρόνια σύμφωνα με μια έκθεση, λέει ότι οι χώρες μέλη θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι υπήρξαν κάποια σφάλματα. Ερώτηση. Διεξήχθη στο Συμβούλιο συζήτηση μεταξύ των 27 ή 28 Υπουργών Οικονομικών για να δείτε τι είδους λύση μπορείτε να δώσετε, να διασφαλίσετε δηλαδή μεγαλύτερη υπευθυνότητα των αρχών των χωρών μελών ώστε να αποφευθούν οι ε, συστάσεις οι δυνατών. Επανερχόμεθα στο, θέμα της σωστής ε, κοινοποίηση των δεδομένων από τις χώρες μέλη των, ε, των ελεγκτών οι χώρες μέλη. Προκειμένου το Συμβούλιο ζητεί από δεν ξέρω αν απαντώ στην ερώτηση σας. Άλλος κανείς, εσείς κύριε Τσέλερ πάλι. Χρονικά συνδέεται με τη Συμφωνία Κοτονού που λίγη ισχύ στο 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως που κινείται ως ξεχωριστός προϋπολογισμός τάξη μεγέθους χρησιμοποιείται ή μέρη του χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως, ενσωμάτωσή του στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ενδεχομένως με αναφορά σκοπού χρήσεως ότι απαλλαγή. Και τούτη εδώ η ερώτηση δεν συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία απαλλαγής. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως σχετικά είναι ότι σίγουρα θα ενταχθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και πάλι σε βάση πρόταση της Επιτροπής. Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι μόνο η ΕΘΟΝ. Εάν δηλαδή το EDF θα μπει στο, θα σωματωθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, θα παραμείνει εκτό. Η δική μα εθνική βουλγαρική θέση είναι ότι θα θέλαμε να παραμείνει εκτό Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει και τη συνέχιση τη Συμφωνία Κότονου, αυτό είναι ερώτημα. Μπορώ να σας δώσω μια ικανοποιητική απάντηση. Ευχαριστώ. Κλείνω εδώ αυτό το θέμα. Συνάντηση αυτή εδώ. Απαντήσατε με ανοιχτό και ειλικρινές πνεύμα τις ερωτήσεις. Η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών για μας είναι πολύ σημαντική. Είπα και πολλά ήδη, αλλά θα πω λίγα ακόμα, αν δεν έχετε αντίρρηση. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων στοιχείες μας για παράδειγμα βελτίωση των μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες, εργασίες σας τις επόμενες εβδομάδες στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής 2019. Goed, dan eh, Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κάντενμπαχ. Είναι η έκθεση 16 κάθετος 2017 με προγραμματισμό στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, με λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. θα έχουμε και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου εδώ, τον κύριο Γιάννους Βοητσεχόφσκι. Και θα έλεγα ε, με την εισηγήτρια και τη συμφωνή γνώμη τη να μας κάνει την παρουσίασή του κύριο Βοητσεχόφσκι για να αρχίσουμε. Ευχαριστώ και πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία το είπατε το όνομά μου. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να σας παρουσιάσω την ε, ειδική έκθεση που έχει ως ε, ε, τίτλο προγραμματισμός αγροτικής ανάπτυξης. Λιγότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Έχω και μια σύντομη παρουσίαση, αν καταστεί δυνατόν να προβληθούν οι διαφάνειες. Πατώ το κουμπί, θα δούμε. Ας περιμένουμε μια στιγμή να δούμε. Λυπούμε για το πρόβλημα, λέει ο κ. Βοητσεχόφσκι. Θα εμφανιστούν τώρα. Μην ανησυχείτε κ. Βοητσεχόφσκι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μου φαίνεται ότι είναι εντάξει τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν γνωρίζετε ότι η πολιτική αγροτικής ή μάλλον ε, ε, ναι, αγροτικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 7 χρόνια της δημοσιονομικής περίοδου δαπανήθηκαν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε στην εικόνα ποια είναι η αναλογία μεταξύ των δυο στυλών. Το 1 τέταρτο της συνολικής δαπάνης για την αγροτική, ε, της αγροτικής, αγροτικής δαπάνης δηλαδή. 14 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. 58 δισεκατομμύρια ευρώ για την γεωργία 14 για ε, άμεσες πληρωμές, 4 για τις αγορές και 14 για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Στην εικόνα αυτή βλέπετε την κατανομή με τις βασικές χώρες που ωφελούνται, Γαλλία, Ιταλία, 11% και οι δύο, Γερμανία 10%, Πολωνία 9%, Ρουμανία 8%. Ε, είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι από τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης. Πάντως, έχουμε 118 RDP project δηλαδή για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτά οργανώνονται από τις χώρες μέλη στο επίπεδο χωρών μελών σε χώρες όπως ε, Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα σε ορισμένες χώρες στο επίπεδο πλέον των περιφερειών όπως στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή και στην Ισπανία. Εξετάσαμε 10 RDP σε Πολωνία, Ρουμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία στην Βαλονία του Βελγίου, στη Βάδη Βιρτεμβέρη της Γερμανίας, περιφέρειες αυτές τώρα, Λαριόχα στην Ισπανία, Καμπανία στην Ιταλία και δύο από τα RDP έγιναν από την ε, Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγγλία και στη Δανία. Τώρα, ποια ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο έλεγχος. Ε, το βασικό ερώτημα του ελέγχου ήταν η έμφαση στην απόδοση, απόδοση περιλαμβάνεται στην νομοθετική ρύθμιση. Τα RTP έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Αυτό ήταν το focus on performance. Εκεί ρωτήσαμε πώς διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την διαδικασία του προγράμματος, την προγραμματική διαδικασία. Τώρα ποια είναι τα βασικότερα συμπεράσματα. Τα επίσημα συμπεράσματά μας είναι ότι τα RDP, τα project δηλαδή, ήταν πολύ γενικά, πολύ μακροσκελή και περίπλοκα. Η προγραμματική διαδικασία ήταν υπερβολικά μακρά και αυτή. Τα δε RDP ήταν ανεπαρκώς απέδιδαν ανεπαρκή έμφαση στα αποτελέσματα. Ας πούμε τώρα λιγότερο επίσημα θα μπορούσα να πω ότι τα βασικά συμπεράσματα είναι τέσσερις φορές το L. Έχουμε δηλαδή τα RDP που ήταν too large, πολύ ευραία, too long, πολύ μακρές προγραμματικές διαδικασίες, too late, πολύ καθυστερημένες και too less, πολύ λίγο δηλαδή, στοχευμένα σε αποτελέσματα. Γιατί λέμε too large, πολύ ευραία. Σας δείχνω μια εικόνα τώρα σε, αυτή την, ε, σε αυτό τον πίνακα καλύτερα βλέπετε πόσο ευραία ήταν αυτά τα RDP, Rural Development Projects. Μια στιγμή με συγχωρείτε. Βλέπετε στον πίνακα ότι στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο 2007 έως 2013 το μέσο μέγεθος των RDP ήταν 459 σελίδες. Το μεγαλύτερο RDP εκείνη την περίοδο ήταν στην Βάδη Βιρτεμβέργη πάνω από 700 σελίδες περιφέρεια της Γερμανίας. Και το πιο μικρό, το πιο σύντομο δηλαδή, ήταν στην Αυστρία, 370 σελίδες. Τώρα, στην περίοδο 2004 έως 20, το μέσο μέγεθος των RDP ήταν 781 σελίδες. Στην Ελλάδα μάλιστα πάνω από 1000 σελίδες. Μόνο στην Ιρλανδία το RDP ήταν μικρότερο κατά μία σελίδα από το προηγούμενο, από την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή 456 σελίδες αντί 457 στην προηγούμενη περίοδο. Γενικά μιλώντας, κάθε RDP έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο, πολύ μακροσκελέστερο από πριν. Κατά τη γνώμη μας, τα έγγραφα αυτά είναι υπερβολικά μακροσκελή και υπερβολικά περίπλοκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί υπερβολικά πολλά από τις χώρες μέλη. Και μετά από πολλές συζητήσεις για την απλούστευση της κοινή αγροτικής πολιτικής, εγώ τα θυμούμαι αυτά και εδώ μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε συζητήσει αυτά στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ ότι χρειαζόμαστε απλούστευση. Σήμερα η κόπα κοζεκά, η οργάνωση των αγροτών, βγαίνει και κάνει επίσημη δήλωση ότι η απλούστευση της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι απόλυτα αναγκαία. Σε αυτά τα RDP, ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε. Έχουν γίνει πιο περίπλοκα τα προγράμματα δηλαδή ε, της ε, αγροτικής ανάπτυξης έχουν γίνει πιο περίπλοκα και πολύ δυσνόητα για τους Γιώργους. Ίσως έχουν κάποια, κάποιο ενδιαφέρον για πανεπιστημιακές μελέτες, αλλά όχι για τους απλούς αγρότες. Αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα. Το επόμενο που λέμε είναι ότι τα RDP είναι, ή μάλλον η προγραμματική διαδικασία είναι υπερβολικά μακρά. Εδώ στο γράφημα που σας δείχνω, σας δείχνουμε πόσο μακρά ήταν αυτή η προγραμματική διαδικασία. Δηλαδή είναι της τάξης περίπου του ενός έτους, λίγο λιγότερο, 11,2 μήνες η μέση διάρκεια. Ορισμένα προετοιμάστηκαν ταχύτερα, άρα χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο. Άρα, για τη γνώμη μας είναι υπερβολικά μακρές οι περίοδοι αυτές. Χάσαμε πολύ χρόνο δηλαδή. Τώρα το επόμενο συμπέρασμα είναι ότι τα RDP εγκρίθηκαν με υπερβολική καθυστέρηση. Υπερβολικά αργά. Είναι καλό το χρονικό αυτό σημείο που είμαστε τώρα να το συζητήσουμε αυτά γιατί είμαστε στην ίδια περίοδο που ήμασταν το 2004, το 2011 στην αρχή δηλαδή τη συζητήσεω για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Ε, κοιτάξτε λίγο το άνω μέρος της εικόνας, της, ε, του πίνακα, λέμε ποια ήταν η κατάσταση 2007 έως 2013. Η πρώτη πρόταση της Κομισιόν τον Ιούλιο του 2004 Κανονισμό του Συμβουλίου την εποχή εκείνη που ήταν ο μόνο νομοθέτης με, με γνωμοδότηση μάλλον του Κοινοβουλίου ε, ο κανονισμό του Συμβουλίου εγκρίθηκε το 2005 το 2006 ήταν, έτοιμη και, ήταν έτοιμος και ο κανονισμός εφαρμογής το 2007 που ήταν ο πρώτος χρόνος, το πρώτο έτος δηλαδή της ε, χρηματοδοτικής περίοδου, όλα ήταν έτοιμα. Σε τούτην εδώ, τη χρηματοδοτική περίοδο, το 2011 κατατίθεται η πρόταση της Κομισιόν, τον Οκτώβριο του 2011, ο κανονισμός που είναι τώρα πια Συμβουλίου και Κοινοβουλίου εγκρίνεται τέλη 2013 στις 17 12 για να είμαι ακριβής οι εκτελεστικοί κανονισμοί εγκρίνονται από την Επιτροπή το 2014. Άρα με καθυστέρηση συγκριτικά με παλαιότερα, με την προηγούμενη φορά και στο επόμενο γράφημα βλέπουμε τις ε, συνέπειες στην πράξη της που έχει αρχίσει η δημοσιονομική προοπτική είναι μόλις της τάξης του 21%. 79% δεν έχει απορροφηθεί δημοσιονομικής ε, περίοδου, το, ο μέσος όρος απορρόφησης ήταν 29%. Ίσως να σας ενδιαφέρει και ο επόμενος πίνακα αγροτική πολιτική και καινούργια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Πότε θα εγκριθούν. Εάν εγκριθούν μετά το 2019 να βάλουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος για να γίνει αποτελεσματικότερη χρήση των χρημάτων χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι των πολιτικών της συστάσεις μας. Νομίζω η πιο σημαντική που είναι ας πούμε στο διατακτικό της έκθεσής μας λέμε τα τρία θεσμικά όργανα και να κάνουν μια σε βάθος επανεξέταση πριν να θεσπίσουν τους συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς ενδιαφέρον. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την ε, κυρία Κάντενμπαχ. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και ιδίω οι κύριοι συνεισηγητές Νοβακόφ Φλάναγκαν και, και ο Μάριο Μπίλιτσεφ, ο οποίο είναι ε, γενικό διευθυντή τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Θα τον παρακαλέσω λοιπόν να απαντήσει στο τέλος εάν προκύψουν ερωτήματα στη διάρκεια τη συζήτηση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάντενμπαχ. Μετά θα ακούσουμε τους άλλους ομιλητέ Κάντε. Σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλούτσεφ από την Κομισιόν και μετά θα έχουμε το γύρο. Το λόγο, α αρχίσουμε τους και οδείς Ο κύριος Νόβακοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανάπτυξη τη υπαίθρου, η αγροτική ανάπτυξη, γίνεται όλο και πιο σημαντική για περισσότερου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο περνάει ο καιρό. Δεδομένη τη φύση του προγράμματο και του είδου των δικαιούχων, πρέπει να το προσαρμόσουμε έτσι ώστε οι δικαιούχοι θα κατανοούν την φιλοσοφία και τη συλλογιστική πίσω από τις δωρεές. Διότι όταν συναντούμε πολίτες από αυτές τις περιοχές, έχουμε την εντύπωση ότι οι περισσότεροι προτιμούν να πάνε στην τράπεζα και να πάρουν ένα δάνειο και να το αποπληρώσουν με τόκο, παρά να έχουν να κάνουν με συμβουλευτική, με consultants και να ακολουθούν περίπλοκες και μακροχρονοβόρες διαδικασίες. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ομάδα δικαιούχων που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου. Άρα μάλλον πρέπει να αλλάξουμε εμείς την διαδικασία και όχι να προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο περίπλοκο. Λέγοντας το αυτό, Δεν προσπαθώ να είμαι απλώς επικριτικός ε, χωρίς αίτιο. Απλώς πρέπει να θέσουμε ένα όριο και να αντλήσουμε διδάγματα από την προηγούμενη περίοδο. Να είμαστε βέβαιοι ότι την επόμενη φορά, εάν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για τη συνοχή και την ανάπτυξη της επέθρου συγκεκριμένα, να φροντίσουμε να προωθηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε ένας δικαιούχος να είναι ουσιαστικά πρεσβευτής υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ αυτών των προγραμμάτων. Ιδάλλως, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε εμείς οι ίδιοι, που νομίζω είμαστε καλύτεροι φίλοι των δικαιούχων εδώ στην Επιτροπή μας, ούτε οι ίδιοι δικαιούχοι, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε αρκετό χρόνο, όχι για μια επανάσταση, αλλά για κάποιο είδους εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της ανάπτυξης της υπαίθρου για το 2021-2027. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βοηθοκόφσκι, το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου για αυτή την έκθεση υψηλής ποιότητας που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, νομίζω πρέπει να προβάλλουμε αυτή τη δουλειά, να ευαισθητοποιήσουμε για το τι έχει επιτευχθεί ως τώρα. Παρόλο που κάποιες φορές είναι κάπως περίπλοκα όσα γίνονται, τουλάχιστον τα αποτελέσματα είναι σημαντικά στην πράξη. Και καλό είναι αυτό να προβάλλεται. Πρόεδρος, ο κύριος Φλάναντον. Ευχαριστώ. Όπως λένε, η πληροφορία είναι εξουσία και οι πληροφορίε που μας δώσατε είναι σαφώ πολύ δυνατέ για να τις αξιοποιήσουμε και να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε το επόμενο διάστημα προγραμματισμού της ΚΑΠ. Εδώ κοιτάζουμε τα ποσοστά απορρόφησης, πρόσληψης όπως το ονομάσατε και από τη δική μου τη χώρα, την Ιρλανδία, βλέπουμε πως περάσαμε από το ποσοστά του 52% σε 38%. Το μόνο που με εκπλήσει είναι ότι δεν έπεσε και περισσότερο το ποσοστό. Διότι από ένα περίπλοκο πρόγραμμα πήγαμε σε ένα ακόμη περιπλοκότερο. Αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον θα ήταν ένα παρόμοιο γράφημα με το 52 και το 38% και το 43% και 48%. Το 52% με συγχωρείτε, το 38% πρόσληψη στην Ιρλανδία και άλλες χώρες να αναλύεται στα ποσά που πραγματικά πήγαν στα χέρια των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Διότι ενώ το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν περίπλοκο και είχαν παραπονεθεί οι δικαιούχοι, τουλάχιστον τους έδινε κάποια χρήματα στο τέλος. Σε αυτό το πρόγραμμα όχι μόνο είναι περίπλοκη διαδικασία, αλλά εξαιτία του περίπλοκου χαρακτήρα το ποσό της χρηματοδότησης τελικά που παίρνει στα χέρια του ο Γεωργός και ο κτηνοτρόφους ουσιαστικά δεν αφήνει τίποτα. Ξέρω ανθρώπους που ανησυχούν για το περιβάλλον, αλλά ανησυχούν και για το πώς θα ε, θρέψουν την οικογένειά τους. Εάν λοιπόν το μόνο που έχουμε να τους δώσουμε είναι ένα πονοκέφαλο, ε, και να έχουν τραβήξει τα μαλλιά τους μέχρι να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Δεν μάθαμε τίποτα το προηγούμενο πρόγραμμα. Λοιπόν, ο κόσμος δεν θα θέλει να συμμετάσχει αν δεν βάλει κάτι και στην τσέπη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό και ως προς τα προγράμματα που βασίζονται στις επιδόσεις και την... Ε, ε, τον ορισμό στόχων σε εθνικό επίπεδο. Καλή ιδέα, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν γελία χαμηλού στόχου στα κράτη-μέλη και μετά να λένε ήρθαμε και πήγαμε και καλύτερα από το στόχο που είχαμε θέσει, να μην ε, το αφήσουμε και αυτό ανεξάρτητο. Όπου συμμετείχα σε τέτοια προγράμματα, πώ έχω καταντήσει στο τρικοτό τη κεφαλή μου. Ε, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορώ παρά να. Παρα... Ε, δαπανήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό είναι ε, ένα πόρισμα του ελεκτικού συνεδρίου εδώ. Φαίνεται ότι τα μισά από αυτά τα χρήματα δεν ταπανήθηκαν. Ποσά από την επόμενη χρονιά, ποσά που δεν απορροφήθηκαν για, να τα, για τις δαπάνες τις φετινές. Φαίνεται να υπάρχουν ε, τεράστιες δαπάνες ε, και διαχειριστές ε, βγάζουν από αυτά ένα μισθό. Το ελεγκτικό συνέδριο καλό αυτό να μας δώσει και ένα σχετικό ποσοστό. Αυτοί οι πτυχιούχοι πανεγαλώνουν με το ψυχοτό της κεφαλής σας σίγουρα, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να πει και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είμαι μέλο ε, μέλος της Επιτροπής αλλά μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, με προσεκαλείστε σε αυτή τη συζήτηση. Έφτασα λίγο αργά γιατί μου σε άλλη συνεδρία, σε μια άλλη επιτροπή. Θέλω όμως να κάνω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα Ενδιαφέρον μου φάνηκε. Ιδίω στην περίπτωση της Ισπανίας βλέπω 13%. προκάλλει την προσοχή. Έχω μια ερώτηση προς την ε, Κομισιόν. Αν έχετε αξιολογήσει την εξή παράμετρο. Προγράμματα ανάπτυξης. Το ένα είναι το εθνικό και τα 17 είναι περιφερειακά. Για να κρίνεται αν η εφαρμογή ήταν καλή ή κακή. Είναι ένα θέμα που αφορά την... Ε, δεν ήρθα από την αρχή συζήτηση, δεν ξέρω αν το αναφέρατε και στο συγγνώμη αν το αναφέρατε. Ο δεύτερος πυλώνας συγχρηματοδοτείται το γεγονό ότι και οι περιφέρειες αλλά και οι χώρε δεν είναι όλε στην ίδια κατάσταση. Άλλε έχουν περισσότερου πόρου, άλλε έχουν λιγότερου, περιφέρειες έχουν λιγότερου κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό να προηγείται και μετά να δρομολογούνται τα προγράμματα και δεν είναι το ίδιο η χρονιά αυτή με τι προηγούμενε Σηματοδότηση. Προσπαθούν, ε, εμείς προσπαθούμε όμως να εξασφαλίσουμε πόρους αντίθετα στα προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη και από τις περιφέρειες. Και ένα τελευταίο γρήγορα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υφιστάμενο πλαίσιο. Με τη μεταρρύθμιση του 2014 έχουμε και το πίδελτα μέχρι το 2020, αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να τα εγκρίνει σε έφθετο χρόνο και πιο πολύ είναι ενδιαφέρον για το δημοσιονομικό πλαίσιο και λιγότερο για τις ανάγκες ξυγχρονισμού της πολιτικής. Πώς το βλέπετε και ποια είναι η άποψη του ελεγκτικού συνέδριου. Γιατί αυτό είναι δύσκολο και θα σημαδέψει, θα σηματοδοτήσει και το τέλος του κουπί ΔΕΛΤΑΠΕ αλλά και την ανάπτυξη. που στέλνουν και άλλες επιτροπές μέλη τους στην δική μας επιτροπή γιατί αυτό εμπλουτίζει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα στην Κομισιόν και μετά στο Ελεκτικό. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ πρώτος. Επανελήφθη εδώ το ερώτημα, ε, το ζήτημα της πολυπλοκότητας και ιδίω για το τελικό δικαιού, για τους γεωργικούς παραγωγούς. Αναφέρθηκαν συμβουλευτικέ υπηρεσίες. Αν το σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών λειτουργεί καλά, θα είναι πολύ πιο εύκολο και για τους γεωργικούς παραγωγούς να λάβουν τις σχετικές συμβουλές και να αναζητήσουν επιχορηγήσεις και όχι δάνεια. Γενικά όμως η ιδέα είναι να πλούστευση και στο μέλλον αυτό θα είναι στα χέρια των κρατών μελών, δηλαδή να καθορίσουν επακριβώς τι θα είναι πολύπλοκο και τι θα είναι απλό για τον τελικό δικαιούχο. Η παρεμβάση στο μέλλον. Σε αυτή την περίοδο τώρα έχουμε τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης Δεν δυσκολεύουμε τη ζωή των γεωργικών παραγωγών, το είπα και πριν. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να εφαρμόζουμε αυτά που λένε οι κανόνε, η νομοθεσία. Αν λοιπόν πλέον η νομοθεσία περιλαμβάνει μόνο τι βασικέ απαιτήσει, οι παρεμβάσει θα σχεδιάζονται ακόμα του παραγωγών. Έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Φλάναγκαν που μα ενδιαφέρει όλου πολύ εμά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ γελιοδός χαμηλό θα το χαρακτήριζα πεδίο στόχων που καθορίζει και το επίπεδο φιλοδοξίας. Και τώρα επεξεργαζόμαστε τους ειδικού στόχους που θα προσδιορίζονται στην νομοθεσία. Με βάση τους στόχους αυτούς θα έχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο φιλοδοξίας. Επίσης, αυτή τη στιγμή καθορίζουμε και τους δείκτες και μιλούμε για τρεις ομάδες δικτών Impact Result Output. Και μαζί με τα κράτη-μέλη θα καθορίσουμε τα επίπεδα φιλοδοξίας και με βάση αυτούς τους δείκτες τα μελλοντικά σχέδια κοινή γεωργική πολιτική που θα περιλαμβάνουν και τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα θα εγκρίνονται από την Κομισιόν. Άρα αυτό το γελιοδό χαμηλό επίπεδο στόχων που αναφέρατε κι εσεί, δεν θα υφίσταται πλέον, γιατί θα συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου και η Κομισιόν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλλον η γάμα δέλτα μπάτζ θα έπρεπε να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική όμως, αυτό που μπορώ να πω, το είπε και ο κ. Βεσεχόφσκι. Ότι τα τρία τέταρτα των δαπανών γίνονται στον πρώτο πυλώνα. Άρα στον πρώτο πυλώνα δεν έχουμε αυτά τα χαμηλά ποσοστά, έχουμε ψηλότερα ποσοστά. Άρα η κοινωνική πολιτική εκπροσωπείται πολύ καλύτερα στι δαπάνε. Η αγροτική ανάπτυξη, το παραλαμβάνω, δεν μας ανησυχεί. Είναι 25% μέσος όρος. Φυσικά έχουμε ερωτηματικά εδώ και εκεί, σε κάποιες περιφέρειες, σε κάποια κράτη-μέλη. Και στις ετήσιες συναντήσεις που έχουμε για τις αξιολογήσεις και στο πλαίσιο των επιτροπών αξιολόγησης, έχουμε επαφέ με αυτά τα κράτη-μέλη και αυτέ τι περιφέρειε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μα ανησυχούν τα επίπεδα όμω. Και προ το παρόν δεν βλέπουμε κάποιο μεγάλο κίνδυνο, να έχουμε decommitment, οδέσμευση κάποιων κονδυλίων. Χρησιμοποιήσει για την κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία το πρώτο ερώτημα. Άμεση απάντηση. Όχι. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του ότι έχουμε κάποια εθνικά και κάποια περιφερειοποιημένα κράτη-μέλη. Γιατί, να σας δώσω και το παράδειγμα της Γερμανίας, που είναι ομόσπονδο κράτο. Υπάρχουν προγράμματα των κρατηδίων που στις περισσότερες περιπτώσεις πηγαίνουν πολύ καλά και γρήγορα. Σε άλλα κράτη, η Γαλλία έχει περιφέρει. Σε κάποιες περιφέρειες ε, οι δαπάνες επίση προχωρούν πολύ καλά. Στην Ισπανία δεν την ανέφερα, δεν την κατονόμασα την Ισπανία, αλλά ναι, το είπατε κι εσείς, ήταν ε, μία από τις χώρες ε, με χαμηλή απορρόφηση και καθυστερημένη έγκριση. Όταν εγκρίθηκαν τότε τα προγράμματα, ήμουν διευθυντής αρμόδιος για την Ισπανία και μπορώ να σας πω ότι κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια ε, για να εργαστούμε με τους ισπανικούς φορείς και να εγκρίνουμε τα προγράμματα επιτόπου. Είχαμε και πολιτικά προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της χαμηλής απορρόφησης δεν ήθελαν να προχωρήσουν γρήγορα με την έγκριση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Για το δεύτερο πυλώνα και τη συγχρηματοδότηση στην αγροτική ανάπτυξη. Είναι θέμα για τους συνομοθέτες και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις περιφέρειες συνοχής έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε χρηματοδότηση και προπολογισμού. Είναι όμως ένα ζήτημα που υπερβαίνει το δικό μου επίπεδο. Το αν θα υπάρξει δηλαδή χρηματοδότηση στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα προβλήματα της η δυνατότητα, η συγχρηματοδότηση ή να μην υφίσταται ή το ποσοστό τη είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ένα τελευταίο ερώτημα που δεν απευθύνεται τόσο. Πολύ θετικέ του αντιδράσει στην έκθεσή του και θα περάσω στα πολωνικά, αν μου επιτρέπετε. Για την κυρία Κάντεμπαξ, σας ευχαριστώ πολύ ε, είστε εισηγήτρια και σας ευχαριστώ για την θετική σας αντίδραση για τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης. Επίσης ευχαριστούμε για τις ε, παρατηρήσεις που μας κάνατε. Είπατε ότι ε, ενδιαφέρουσες δημοσίευσεις, συγκεκριμένα ένα αναλυτικό κείμενο που συνοψίζει το τι διαπιστώσαμε από διάφορες εκθέσεις που είχαν προηγηθεί, η κατανόηση. Νομίζω ότι από κοινού συνεργαζόμαστε για το κοινό συμφέρον, το οποίο έγκυται στο να προσαρμόσουμε την κοινή αγροτική πολιτική στι μελλοντικέ ανάγκε. Να μην υπάρχουν ιδιαίτερα περίπλοκέ διαδικασίε. να μην χρειάζεται να ε, απευθυνθούν σε κονσάλταντ και συμβούλου. Θα πρέπει ο κάθε πολίτη που δεν είναι γεωργός κειμένων, Γι' αυτό επιδιώκουμε την απλούστευση. Προ τον κύριο Φλάναγκαν, σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρατηρητήσή σας και επίσης και προς τον κύριο Άγγιν. για το τι συμβαίνει ε, στι περιοχέ τη Επέθρου συγκεκριμένα. Αυτό είναι μέρος ε, του προγράμματος εργασιών μας για το 2019. Δηλαδή, μια ανακριμένα στοιχεία για το θέμα. Και προς τον κύριο Άγνιου να πω ότι ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο μας κάνατε μια παρατήρηση. 5% του συνόλου, Πολωνία, ε, πήγε κάποια ποσά από τον δεύτερο πυλώνα στον πρώτο. Ε, μεταφορές που είναι καθόλου εφικτέ. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία από την Ισπανία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και ο έλεγχος για την ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου έδειξε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι ένα πρόβλημα εξόχως πολιτικό. δείχνει πώς λειτουργούν ορισμένα κρατημέλη και πώς ο προγραμματισμός γίνεται είτε σε επίπεδο κεντρικά, είτε σε επίπεδο περιφερειακό και επίπεδο κρατών μελών. Αυτά, Πρόεδρε, και για να ολοκληρώσω, να ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα σήμερα να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας.